Good afternoon. Good afternoon. I reopen. Καλησπέρα. Κυρίσω την έναρξη της συνεδρίασης για να συνεχίσουμε. Ελπίζω να φάγατε καλά. Πριν αρχίσουμε, έχω ένα πρακτικό ζήτημα. Μια παρατήρηση για την οργάνωση. Στα προγράμματά σας τα είδατε ότι θα προσπαθήσουμε σήμερα το απόγευμα να κάνουμε ένα πείραμα για να έχουμε μια πραγματικά διαδραστική συνεδρίαση μεταξύ μας, μεταξύ των βουλευτών. Δηλαδή να μην απευθύνετε ερωτήσεις και να μιλάτε με το πάνελ μόνο, αλλά και μεταξύ σας. Αυτό είναι κάτι που θα αποτελέσει και τη βάση για τις επόμενες συνεδριάσεις. Θέλουμε λοιπόν να προσπαθήσουμε. Αν κάποιοι... Εσείς που είσαστε πίσω-πίσω, Μπορείτε να έρθετε πιο μπροστά. Πάρτε και τα πράγματά σας στην καρτέλα με το όνομά σας για να γεμίσουν οι πρώτες σειρέ εδώ στο εμικύκλιο για να βλεπόμαστε και καλύτερα. Μπορείτε να έρθετε παρακαλώ πιο μπροστά. Πάρτε και τα πράγματά σας, ελάτε μπροστά. Για να είναι έτσι πιο κλειστός ο κύκλος, πιο μικρός. Θα είναι πιο εύκολο, αφού έχουμε ακούσει τους δύο κεντρικούς μας ομιλητές, μετά να συζητήσουμε και μεταξύ μας. Λοιπόν, λίγα λεπτά για να γίνει αυτό. I see some movements, that's good. Βλέπω κάποια κίνηση. Φιλανδία εκεί πίσω. Ελάτε πιο μπροστά. Ελάτε κι εσείς πιο μπροστά παρακαλώ. Ναι, σας βλέπω. If you could cooperate, please, then, uh, because also... Συνεργαστείτε παρακαλώ, γιατί αν θέλουμε να συζητήσουμε με αυτόν τον τρόπο είναι σημαντικό να βλεπόμαστε καλύτερα. Να μπορεί ο πρόεδρος να σας προσέξει αν θέλετε το λόγο κλπ. Γι' αυτό ελάτε πιο μπροστά παρακαλώ.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 back, would you like to move a little bit forward? forward? Εσείς εκεί πίσω μήπως θέλετε να είστε λίγο μπροστά, είστε καλά. Άμα θέλετε να μιλήσετε όμως θα ε, κουνάτε το χέρι σας, χοροπηδάτε να σας δούμε. <laughs> I see the ladies uh, moving. Okay, thank you. Ευχαριστώ. Να προσπαθήσουμε τώρα να προχωρήσουμε. Να δώσω με ιδιαίτερη χαρά το λόγο στον κύριο Τόμας Χάντελ. Αγαπητοί συνάδελφοι, να σας καλωσορίσω στην επόμενη συνεδρίασή μας προσεχή σενάρια για τις επενδύσεις σε μια ανταγωνιστική Ευρώπη, οι δυνατότητες και οι προκλήσεις επειδή βλέπω ότι σας παρακάλεσαν ε, να κινηθείτε ε, θα ήθελα να σας συστήσω τον συνάδελφο κύριο Ντούζενμπεργκ που το γνωρίζουμε είναι πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών εγώ με Τόμας Έντελ είμαι ο πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Θεμάτων είχα την ευκαιρία να προεδρεύσω χθε με τον συνάδελφο Φέρμπερ μερικές παρατηρήσεις τεχνικής φύσης τώρα για τη συνεδρίαση αυτή. Δεν χρειάζεται να μας στέλνετε σημειώματα, απλώς θα σηκώνετε το χέρι σας. Εδώ οι συνάδελφοι στο Προεδρείο θα καταγράφουν τα ονόματά σας, ούτως ώστε να υπάρχει εναλλαγή εθνικών και ευρωβουλευτών. Έχουμε και τις 23 γλώσσες της Ένωσης. Θα έχετε λοιπόν τη δυνατότητα στην επόμενη μια μισή ώρα να συζητήσετε πολλά θέματα. Αυτά για πρακτικά ζητήματα. Οπότε, θέλω να τονίσω ότι σε αυτόν το γύρο συζητήσεων θα ασχοληθούμε με το θέμα της πολιτικής επενδύσεων για τη δημιουργία απασχόλησης και φυσικά και με το θέμα των μελλοντικών επενδύσεων, πώς θα επενδύσουμε στους συμπολίτες μας, στους συμπολίτες που θα πρέπει να είναι οι δημιουργοί της οικονομίας του μέλλοντος. Είναι λοιπόν συναρπαστικό αυτό το καταληκτικό πάνελ. Έχουμε δύο εισηγητές. Χαιρετώ την Λάουρα Φανχέστ που είναι διευθύντρια του Ολλανδικού Γραφείου πολιτικών και οικονομικών αναλύσεων και θα σας παρουσιάσει το θέμα της ε, σε ένα τέταρτο. Ελπίζω να μην είναι πολύ περιοριστικό, αλλά ο χρόνος πάντα μας περιορίζει. Και επίσης έχουμε την Μαρή Κιλινιέμι, που είναι αναπληρώτρια γενική γραμματέας του Οργανισμού Οικονομικής Ανάπτυξης Εργασίας του ΟΣΑ. 10 λεπτά λέει εδώ το σημειωμά μου, αλλά εάν θέλει λίγο περισσότερο χρόνο δεν θα είμαι άκαμπτος. Αυτά. Θέλουμε να κατανείμουμε σε διάφορες φάσεις της συζήτησης και πώς θα προχωρήσουμε μετά θα πει ο συμπρόεδρος μου, κύριος Ντουίζλμπερ. Λοιπόν, να γίνουν οι δύο παρουσιάσεις και μετά θα κάνουμε τη συζήτηση. Πρώτη λοιπόν η κυρία Φανχέιστ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τιμή μου που είμαι εδώ σε μια τόσο μεγάλη αίθουσα συνεδριάσεων. Δεν έχω ξαναμπεί σε τόσο μεγάλη αίθουσα. Λέγομαι Λόρα Φανχέιστ, είμαι διευθύντρια του Γραφείου Ανάλυσης ε, του, ε, του Γραφείου Αναλύσεων για Οικονομικά και Κοινωνικά Θέματα. Θέλουμε να κάνουμε αναλύσεις για διάφορα θέματα και στο εσωτερικό και εκτός της Ολλανδίας. Είμαστε ανεξάρτητος οργανισμός. Θεωρούμε ότι είμαστε σαν την υπηρεσία Google Translate για όσους ασχολούνται με τέτοια θέματα. Θέλουμε να κάνουμε συστάσεις που να είναι και χρήσιμες για τους πολιτικούς και για ε, την ακαδημαϊκή έρευνα. Εμείς κάναμε τις προτάσεις για τα IFI δηλαδή τους ανεξάρτητους ε, δημοσιονομικούς οργανισμούς καθώς και για τις, ε, τα, τα συμβούλια ανταγωνιστικότητας. Να στραφώ τώρα στον σημερινό ρόλο. Το ρόλο των ε, δημοσίων επενδύσεων για την προώθηση των επενδύσεων στην μετα υφεσιακη εποχή. Γιατί υπήρξε ύφεση η ανάπτυξη είναι αρκετά αδύναμη θα έλεγα ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον τεχνικό όρο σαν το σαλιγκάρι 2% περίπου για την Ένωση και 1,7 για την Ευρωζώνη 1,7 έως 1,9 και, και η ανεργία παραμένει υψηλή η μεγάλη ύφεση με την οικονομική κρίση ακόμη έχει τις επιπτώσεις τα σημάδια Υπάρχουν πολλές επιπτώσεις στα νοικοκυριά, στον ιδιωτικό τομέα, πολλά νοικοκυριά αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγασης. Η πολύ βραδία επίλυση των ε, τραπεζικών προβλημάτων έχει να κάνει με τις δυνατότητες δανειοδότησης και φαίνεται ότι έχει επανέλθει η αβεβαιότητα για την πορεία προς το μέλλον. Μήπως όμως αυτή είναι η νέα παγκόσμια κατάσταση την οποία θα πρέπει να συνηθίσουμε ή θα επανέλθουμε σε καλύτερε εποχές και τι μπορεί να κάνει η πολιτική για να μα εμποδίσει σε αυτό. Βεβαίω, ε, αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις ε, έχουν ε, κάνει ό,τι μπορούν. Η νομισματική πολιτική μέσω τη ποσοτικής χαλάρωσης έκανε ό,τι μπορούσε αν και συζητιέται η αποτελεσματικότητα και γίνεται συζήτηση και για το εάν θα πρέπει να κάνει περισσότερα η δημοσιονομική πολιτική. Θα πρέπει να έχουν υπάρξει περισσότερε δημόσιες επενδύσεις, επειδή είναι τόσο χαμηλά τα επιτόκια και διότι θα μπορούσε να υπάρξει μόχλευση του δημόσιου προς τον ιδιωτικό. Λοιπόν, πώς έχουν τα πράγματα. Ποια είναι η κατάσταση των επενδύσεων. Εδώ βλέπετε πώς ε, έχουν εξελιχθεί επενδύσεις από το 1995. Βλέπετε λοιπόν ότι επενδύσεις είναι ένα υπολογίσιμο τμήμα του ΑΕΠ κατά γενικό 22,4 πριν από την κρίση ενώ μετά το 2008 οι επενδύσεις κατέρευσαν. Εδώ βλέπετε στο Euro 15 είναι η κίτρινη. Η Ιαπωνία είναι το κίτρινο. Το, συγγνώμη, η Ιαπωνία είναι το μπλε, οι Ηνωμένες Πολιτείες κόκκινο, η 15 κίτρινο και ο ECD μαύρο. Όλες οι χώρες ε, είχαν προβλήματα, αλλά ορισμένες έχουν ανακάμψει. Με άλλο τρόπο. Δείτε τι γίνεται στην Ιαπωνία. Να δούμε τι είδους επενδύσεις έχουμε. Έχουμε την κίτρινη γραμμή που είναι οι επιχειρηματικές επενδύσεις, ο στεγαστικός τομέας ε, το μπλε και οι δημόσιες επενδύσεις το κόκκινο. Εδώ διαπιστώνουμε ότι οι περισσότερες είναι λοιπόν επιχειρηματικές επενδύσεις. Μετά είναι στεγαστικές και μετά δημόσιες η ροζ γραμμή και βλέπετε ότι έχει αλλάξει ο συσχετισμός οι επενδύσεις ε, για τη στέγαση μειώθηκαν ήδη από το 2006 πριν από την ύφεση ενώ οι επενδύσεις ε, των επιχειρήσεων τα πήγαν καλύτερα αμέσως μετά την κρίση ενώ οι δημόσιες επανήλθαν με πολύ αργότερο ρυθμό για να δούμε γιατί μειώθηκαν οι επενδύσεις βλέπετε πως ε, μειώθηκαν το κίτρινο επιχειρήσεις, πράσινο στέγαση, ροζ δημόσιες. Από την συνολική μείωση ε, στο 2,4% του ΑΕΠ σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο η μείωση είναι 40% ε, για τους άλλους δύο τομείς ενώ για τις δημόσιες μόνο 20%. Δηλαδή μειώθηκαν οι δημόσιες αλλά αργότερα και λιγότερο. Εδώ βλέπετε αυτές τι τις επενδύσεις όπως ήταν παλιότερα. Αλλά τώρα έχουμε και ένα νέο είδος επενδύσεων, έρευνα και ανάπτυξη. Και εδώ βλέπετε πώ έχει εξελιχθεί η έρευνα και ανάπτυξη σε αυτή την περίοδο. Βλέπετε τη σύγκριση μεταξύ 2007 και 2012. Βλέπετε ότι οι επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη δεν υπέστησαν μεγάλες περικοπές. Βλέπετε ότι το πράσινο είναι περισσότερο από το πορτοκαλί. Και θα δείτε συνολικά, ε, ακριβώς πάνω από εκεί που λέει 2007 από κάτω, το μέσο όρο για την Ευρώπη των 15. Τώρα το ερώτημα είναι προς τα πού θα γίνουν οι ιδιωτικές επενδύσεις. Έχουν μειωθεί οι επενδύσεις, κάποιες όμως ανακάμπτουν. Πού θα γίνουν, σε ποιους τομείς. Θα, βοηθήσει, θα βοηθήσουν οι επενδύσεις την ε, ανάπτυξη στον ίδιο βαθμό ή όχι δεν ξέρουμε, αλλά μπορούμε να εικάσουμε τα εξή. Πιστεύουμε ότι οι επενδύσει μπορεί να επανέλθουν σε ένα βέλτιστο επίπεδο, που για αυτές βέβαια, ε, βέλτιστο, που θα είναι χαμηλότερο από την περίοδο πριν την κρίση. Γιατί στο παρελθόν πολλές επενδύσεις γινόταν στο στεγαστικό τομέα, ήταν μια φούσκα του οικονομικού τομέα λοιπόν, δεν θέλουμε να επανέλθουμε σε αυτή. <clears throat> Δεύτερον, η ένταση απόδοσης κεφαλαίων μειώνεται όπως περνάμε από τον κατασκευαστικό κλάδο στις υπηρεσίες και επίσης έχουν μειωθεί και οι τιμές. Για παράδειγμα, οι υπολογιστές και οι τεχνολογίες πληροφορικής είναι φτηνότερες τώρα, άρα θα είναι χαμηλότερο το ποσό που θα επενδυθεί σε αυτές. Και γενικότερα η πτώση του ΑΕΠ θα οδηγήσει σε πτώση των επενδύσεων. Εάν δεν είναι επαρκή ή αργή η ανάκαμψη των επενδύσεων στον ιδιωτικό τομέα, γιατί να μην αυξήσουμε τι δημόσιε επενδύσει. Πολλά επιχειρήματα αναφέρονται. Έχουμε χαμηλά επιτόκια. Γιατί λοιπόν να μην κάνουμε δημόσιε επενδύσει. Και ο φορέα μου λοιπόν έχει μια πιο σφαιρική προσέγγιση. Δεν θα πρέπει να εξετάσουμε τα επιτόκια της Κεντρικής Τράπεζας ε, σε αυτή τη φάση γιατί πρόκειται για επιτόκια χωρίς κίνδυνο. Θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και ένα ποσοστό κινδύνου, ακόμη και αν είναι χαμηλό. Αλλά στην ανάλυση κόστους ε, ωφελήματος βλέπουμε ότι έχει μειωθεί το ποσοστό του επιτοκίου που οφείλεται στην κάλυψη του κινδύνου. Έχει πάει από το 5 στο 4. Αλλά είναι ενδιαφέρον και αυτό το επιτόκιο. Χαμηλότερο από παλιά. Άλλο επιχείρημα υπέρ δημοσίων επενδύσεων, ότι θα δαπανηθούν τα χρήματα αυτά. Υπάρχει λιγότερος κίνδυνος ότι η χρηματοδότηση λίγα αποταμίευση. Αν γίνει συντονισμένη προσπάθεια, όλες αυτές οι επενδύσεις θα είναι ε, και θα έχουν και ένα βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα στην κατανάλωση, το εκκινσιανό αποτέλεσμα ας πούμε. Όμως ως οικονομολόγος και όπως ξέρετε οι οικονομολόγοι πάντα τονίζουν ότι έχουν δύο μεριές πάντα τα επιχειρήματα τους. Λένε από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά. Πρέπει να σκεφτούμε και τους κινδύνους. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Οι επενδύσεις γίνονται σε οδούς, σιδηρόδρομους, γέφυρες. Αν δεν είναι επενδύσεις ε, στην εκπαίδευση που θα ήταν επίσης χρήσιμες. Βέβαια δεν είναι επένδυση με την ε, αυστηρή έννοια, δεν το επιτρέπουν οι υπεύθυνοι των στατιστικών υπηρεσιών να τη θεωρήσουμε επενδύσεις. Αλλά εάν πρέπει ένας δημόσιος οργανισμός, το δημόσιο, να εξετάσει πού θα επενδύσει, η εκπαίδευση έχει πολύ καλή απόδοση. Ένα ευρώ στην εκπαίδευση οδηγεί σε 8-10 ευρώ στο μελλοντικό εισόδημα του μαθητή. Άρα, καλή απόδοση. Άλλο επιχείρημα. Υπάρχει μια λύση που να είναι κατάλληλη για όλες τις χώρες. Όλες οι χώρες πρέπει να κάνουν παραπάνω δημόσιες επενδύσεις και είναι όλες σε να το κάνουν. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες δυνατότητες. Ορισμένα κράτη-μέλη έχουν περιορισμένο περιθώριο ελιγμού. Δεν θέλουν, όλες, ε, δεν θέλουν χρηματαγορές να χρηματοδοτήσουν όλες τις δημόσιες επενδύσεις. Και ορισμένες χώρες πρέπει να κάνουν ακόμη αρκετά για να σεβαστούν τις υποχρεώσεις του Συμφώνου Σταθερότητας. Να σας δείξω μερικές εικόνες τώρα από την Ολλανδία. Με συγχωρείτε που ασχολούμαι με τη χώρα μου. Δείτε πώς έχουν οι δαπάνες για τις υποδομές μεταφορών ε, ως ποσοστό του ΑΕΠ. Θα μπορούσατε να πείτε ότι δεν κάνει και τόσο πολλά η Ολλανδία σε σχέση με άλλες χώρες. Θα μπορούσε να κάνει περισσότερα. Αλλά δείτε τώρα εδώ τι γίνεται. Εδώ βλέπετε αριστερά έχω, εδώ έχουμε την πυκνότητα υποδομών μεταφορών. Γιατί υπάρχει λόγος. Γιατί έχουμε ήδη πυκνό δίκτυο. Όχι μόνο έχουμε πολλούς δρόμους. Οι πολίτες είναι ικανοποιημένοι από αυτό. Γιατί αν δείτε εδώ τι λέει δεξιά Βλέπετε ότι η Ολλανδία είναι μεταξύ των πρώτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευρά ε, βαθμολόγηση για την ποιότητα των ε, υποδομών μεταφορών. Άρα, ναι μεν τα νούμερα σου λένε θα μπορούσε να δαπανίσει κι άλλα, αλλά άμα δει πώ είναι η κατάσταση, δεν θα έβγαζε το ίδιο συμπέρασμα. Και το ίδιο, ίδιο και αν δούμε τις δαπάνες. Όλοι βεβαίως, όλες τις χώρες υπάρχουν δαπάνες δημόσιας και ιδιωτικά σε εκπαίδευση. Εδώ βλέπετε τι δαπάνε αναμαθητή. Αν δείτε αυτό το γράφημα θα λέγατε δεν είναι και τόσο πολλά αυτά που δαπανάει η Ολλανδία που είναι η μπλε στήλη. Αλλά δεν είναι τόσο κακά τα αποτελέσματα γιατί άμα δείτε εδώ τη βαθμολόγηση της Ολλανδίας για την ποιότητα τη εκπαίδευσή τη με βάση τι ε, μελέτε τη πίζα, θα δείτε ότι είμαστε από του καλύτερους. Άρα το θέμα δεν είναι μόνο που μπορώ να ξοδέψω περισσότερα, αλλά και το πώς θα ξοδέψω περισσότερα. Γιατί όπως ξέρετε, οι δημόσιες επενδύσεις ε, χρειάζονται πολύ χρόνο για να υλοποιηθούν. Στην Ολλανδία είναι 7 χρόνια, ίσως να είναι υπερβολικό. Αλλά αυτό σημαίνει ότι αν πω ότι σήμερα θα φτιάξω έναν δρόμο, δεν σημαίνει ότι αύριο θα τον έχεις. Υπάρχουν λοιπόν λόγοι για δημόσιες επενδύσεις αλλά υπάρχουν και προσκόμματα. Σε ενωσιακό επίπεδο το σχέδιο Juncker προσπαθεί να λύσει αυτά τα προβλήματα. Ορισμένες χώρες έχουν περισσότερο περιθώριο να δαπανίσουν, ορισμένες χώρες έχουν περισσότερες ανάγκες δημοσίων επενδύσεων και εδώ έχει η συγχρηματοδότηση το ρόλο της να παίξει. Επειδή είναι ενωσιακό σχέδιο, πρέπει να λάβει υπόψη και εξωτερικούς παράγοντες, αλλά ακόμη και το σχέδιο Juncker δεν είναι εύκολο να εκτελεστεί από πλευράς διοικητικής. Θα τα καταφέρει λοιπόν να εφαρμοστεί γρήγορα. Θα το δούμε. Και τέλος, ελπίζω να μην ε, ξεπέρασα το χρόνο μου. Δεν είναι μόνο οι επενδύσεις που θα βοηθήσουν να έχουμε ανάπτυξη. Βεβαίως οι δημόσιες επενδύσεις μπορούν να παίξουν το ρόλο τους, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορείς να κάνεις. Για παράδειγμα, να επενδύσεις στην καινοτομία και την εκπαίδευση, όπως είπα, Επίσης μπορεί να κάνεις ε, διαθροτικές μεταρρυθμίσεις. Και ακόμη και εδώ υπάρχουν πολλά περιθώρια ωφελημάτων. Μελέτες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έχουν υπολογίσει ότι αν μειωθούν οι ρυθμίσεις και το ρυθμιστικό πλαίσιο και αν γίνουν και μεταρρυθμίσεις στον τομέα των εργασιακών σχέσεων και λέγεται λοιπόν ότι μέσω αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου μπορείς να έχεις μια αύξηση 5-6% του ΑΕΠ και η μεταρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων μπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ κατά 3%. Συνοψίζω, είναι ιδιαίτερα αργή η ανάπτυξη και παραμένει υψηλή η ανεργία και μειώνεται με πολύ χαμηλό ρυθμό. Οι δημόσιε επενδύσει μπορούν να παίξουν ρόλο, αλλά πρέπει επίση να επενδύσουμε και στην εκπαίδευση και να μην αγνοήσουμε τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φανχέιστ. Η κυρία Κιβινιέμι έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σα. Και ευχαριστώ και την Ολλανδία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που οργάνωσαν στη συνάντηση αυτή. Το θέμα έχει επιλεχθεί πολύ καλά και οι κάτω χώρες έχουν κάνει πολλά για αυτό το θέμα και ο ΩΣΑ πέρυσι όταν ο Πρωθυπουργό ε, επισκέφθηκε το Γενικό Διευθυντή μας είπε ότι είχε τρεις προτεραιότητες στην Προεδρία του MCM και ήταν επενδύσεις, επενδύσεις και επενδύσεις. Με όποια σειρά βάλτε το. Με όποια σειρά θέλετε βάλτε το. Αλλά ακριβώ περί αυτού πρόκειται. Και η δουλειά που κάνετε είναι γνωστή στον ΩΣΑ. Τώρα, θα σας δείξω αυτή την πρώτη διαφάνεια. Δεν σας δίνει κάποια πληροφορία. Εδώ όμως η κυρία Φανχέ στη δικιά της παρουσίαση ήδη σας έδωσε μια καλή εικόνα του που βρισκόμαστε σήμερα και δεν έχω πολλά να προσθέσω σε αυτό. Όσον αφορά την ανάπτυξη, θα έχουμε την δεύτερη επισκόπησή μας του χρόνου. Ε, συγγνώμη, αύριο, οπότε δεν μπορώ να σας δώσω σήμερα τα στοιχεία, αλλά εκπλήξεις δεν θα υπάρχουν. Η ανάπτυξη δεν έχει φτάσει ακόμα στα επίπεδα τα οποία θα επιθυμούσαμε και χρειάζονται. Πέρυσι δεν ήταν καλά, ίσως φέτος να είναι λίγο καλύτερα τα στοιχεία. Πάντως, αν δείτε τα στοιχεία για τις επενδύσεις, εδώ αριστερά, στον ΩΣΑ, οι επενδύσεις έχουν επανέλθει σε επίπεδο που ήταν στην αρχή της κρίσης, συνολικά. Και αν δείτε την Ευρωζώνη, οι επενδύσεις είναι 10% πιο κάτω και για μερικές περιπτώσεις σε μερικές χώρες είναι πολύ πιο χαμηλά. Άρα εδώ πολλά πρέπει να γίνουν για να έχουμε περισσότερες επενδύσεις που είναι αναγκαίες άμα θέλουμε ανάπτυξη. Εδώ, σε αυτή τη διαφάνεια, βλέπετε την κατάσταση των επιχειρήσεων. Δεν επενδύουν, είναι απρόθυμες και σε μερικές περιπτώσεις δεν είναι σε θέση να επενδύσουν, δεν μπορούν. Αυτή η διαφάνεια βασίζεται σε στοιχεία που έχουμε από το 2015 από την επισκόπηση για το επιχειρηματικό κλίμα. Γιατί δεν γίνονται επενδύσεις. Είναι θέμα της εσωτερικής και παγκόσμιας ζήτησης, είναι η αβεβαιότητα σε πολιτικό επίπεδο και είναι και ρυθμιστικά εμπόδια που εμποδίζουν επενδύσεις υψηλών επιδόσεων και αποδόσεων. Βέβαια, υπάρχουν και οικονομικοί περιορισμοί πάντα. Σε πολλές χώρες της Ευρωζώνης, ιδιαίτερα σε εκείνες που χτυπήθηκαν περισσότερο από την κρίση, τα δάνεια προσφέρονται με τέτοιο τρόπο που εμποδίζουν την ε, απόδοση στις τράπεζες. Δεν πληρώνονται έπειτα υπάρχουν περιορισμοί και από τα μέτρα τα οποία τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν ε, το αποτέλεσμά τους και οι τράπεζες δεν δανείζουν παραπάνω. Συνεπώς, το πρώτο που θα ήθελα να πω και το βλέπετε εδώ σε αυτή τη διαφάνεια, κυρίως όταν σκεφτόμαστε τις προπτικές για, για βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη, Ερχόμαστε στο θέμα της ζήτησης, πώς θα αυξηθεί η ζήτηση. Εδώ βλέπετε τις εκτιμήσεις μας. Όταν όλες οι χώρες ΟΣΑ παίρνουν μέτρα για να αυξήσουν τις επενδύσεις κατά μισή μονάδα του ΑΕΠ τους, τι επιπτώσεις έχει αυτό στην ανάπτυξη του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι εφικτό με κοινή δράση να αυξήσουμε το ΑΕΠ περισσότερο, να παρεύουμε στο χρέος και άρα να έχουμε ωφέλη. Επίσης μετρήσαμε η Ευρωζώνη αν έκανε κάτι από μόνη της, χωρίς άλλες χώρες όσα τότε και τότε τα αποτελέσματα θα ήταν θετικά. Όχι βέβαια όπως στην περίπτωση που όλες οι χώρες όσα συμμετείχαν στην προσπάθεια, αλλά παρόλα αυτά θα υπήρχαν ωφέλη. Τα προγράμματα ποιότητας τώρα πρέπει όντως να είναι ποιότητας και πρέπει να υπάρχουν και διαρθρωτικά μέτρα συγχρόνως. Και ερχόμαστε εδώ. Μία από τις συστάσεις μας κλειδί είναι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσει. Είναι αναγκαίες. Και εδώ βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια ότι ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων αυτών είναι χαμηλός στην Ευρωζώνη. Χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις καλά στοχευμένες που να βοηθήσουν την ενίσχυση της παραγωγικότητας, την απασχόληση και προοπτικές ανάπτυξης μακροπρόθεσμα. Πρέπει να βελτιωθεί το περιβάλλον και να διευκολυνθεί η δυνατότητα νέων δραστηριότητων και στο εσωτερικό και διασυνοριακά. Χρειάζονται λοιπόν μέτρα υπέρ της αγοράς εργασίας και της παραγωγής. Πρέπει να κοιτάξετε επίσης και τις στρατηγικές σας για την καινοτομία την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Τώρα για αυτό το περιβάλλον που λέγαμε, πώς θα γίνει πιο ευνοϊκό. Υπάρχει ένα πλαίσιο πολιτική στον ΩΣΑ υπέρ των επενδύσεων που προσφέρει έναν χάρτη πορείας. Με το εργαλείο αυτό οι χώρες μπορούν να αναπτύξουν τα δικά τους συστήματα με περισσότερο διαφανή τρόπο έτσι ώστε να είναι πιο προβλέψιμο το μέλλον και το επιχειρησιακό περιβάλλον για τις επενδύσεις. Έτσι οι χώρες μπορούν να προωθήσουν στην πράξη τις επενδύσεις. Σας ενθαρρύνω λοιπόν να το χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο που διαθέτουμε. Έρχομαι τώρα στις ρυθμίσεις. Εδώ, σε αυτή τη διαφάνεια, βλέπετε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Διαφορές μεταξύ των χωρών όσον αφορά τις ρυθμίσεις τους. Σε κάποιους τομείς υπάρχουν επενδύσεις σε δίκτυο όπως είναι το ενεργειακό, οι μεταφορές και τηλεπικοινωνίες. Οι περίπλοκες ρυθμιστικές διαδικασίες επηρεάζουν και τις εσωτερικές επενδύσεις. Πολλές φορές υπάρχουν εμπόδια για να επενδύσει κανείς στο εξωτερικό. Είναι όμως ενδιαφέρον γιατί δεν πρόκειται μόνο για τους περιορισμούς εξαιτία των ε, ρυθμίσεων, δεν φταίει μόνο αυτό για τον περιορισμό των επενδύσεων. Φταίει το γεγονός ότι είναι διαφορετικές οι ρυθμίσεις αυτές μεταξύ των χωρών. Όσα λοιπόν όσο από τη δουλειά του έχει δείξει ότι υπάρχει αυτή η διαφορά και έτσι εμποδίζονται οι επενδύσεις και το εμπόριο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να λάβει υπόψη της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται δηλαδή πρόοδος προς ε, την κατεύθυνση της εναρμόνισης στην Ευρώπη. Μετρήσαμε επίσης και υπολογίσαμε ότι με 20% μείωση τις διαφορές ε, στην ε, ρύθμιση μεταξύ των χωρών μελών θα μπορούσε να αυξήσει με 13 έως 20% την αύξηση των επενδύσεων και του εμπορίου. Άρα λοιπόν μπορεί να λειτουργήσει σαν μοχλός. Σε αυτή την επόμενη διαφάνεια συνοψίζουμε τις συστάσεις του ΟΣΑ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι από τρεις μελέτες που έχουμε κάνει και θα πάνε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες μέλη. Είναι στις τακτικές εκθέσεις που κάνουμε κάθε χρόνο. Το Μάιο θα τα πάρετε. για το επενδυτικό σχέδιο της Ευρώπης. Το υποστηρίζουμε ενθουσιοδός. Προχωρήστε σε αυτό λοιπόν. Όταν θα έχει προχωρήσει, θα ωφελήσει ολόκληρη την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θα αυξηθούν οι επενδύσεις σημαντικά. Χρειάζεται όμως η αποδοχή υψηλότερων κινδύνων. Αν θέλουμε να πετύχουμε το στόχο των 350 δισεκατομμυρίων σε τρία χρόνια. Υψηλότερος κίνδυνος από ό,τι δέχονται μέχρι τώρα τα περισσότερα επενδυτικά σχέδια. Δεν πρόκειται όμως μόνο για τη ρύθμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. πρέπει να κοιτάξουμε τι γίνεται και πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όσα λοιπόν παίζει ενεργό ρόλο στο θεματολόγιο του G20 και εντοπίζει τις προκλήσεις που υπάρχουν όσον αφορά τις στρατηγικές της επενδυτικές διαφόρων χωρών. Μια μεγάλη πρόκληση είναι οι θεσμικοί επενδυτές να είναι σταθεροί και να συνεχίζουν και να υποστηρίζουν με επενδύσεις τις διαρθρωτικές αλλαγές. Και αυτό είναι στην καρδιά του προγράμματος του ΟΣΑ. Και αυτό προσπαθούμε να προσφέρουμε στις χώρες μέλη. Πώς να ενισχυθούν οι επενδύσεις των θεσμικών επενδυτών. Τέλος, ποιο είναι το μήνυμά μου. Αυτό που πραγματικά χρειάζεται είναι δημοσιονομικά εργαλεία για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ζήτησης και μεταρρυθμίσεις για να έρθουν τα εμπόδια και χρειάζονται μακροχρόνιες επενδύσεις. Κυρίως όταν πρόκειται για τις ευρωπαϊκές χώρες που, όπου χρειάζονται χρηματοδότηση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί εκείνοι που βρισκόμαστε πίσω σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα άλλο στοιχείο είναι η πολιτική βεβαιότητα. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Συνεπώς, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η άποψη τόσα για το τι πρέπει να γίνει και από εκεί πέρα είμαι στη διάθεσή σας για συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε λοιπόν δύο παρουσιάσεις, δύο απόψεις και τώρα έχετε το λόγο για να μιλήσετε εσείς οι εκπρόσωποι και στις δύο παρουσιάσεις εν μέρη είχαμε την ανάλυση του προβλήματος και μια εικόνα της κατάστασης που έχουμε σήμερα και το γεγονός ότι έχουμε πολύ βραδία ανάπτυξη με ρυθμούς χελώνας αν μπορώ να χρησιμοποιήσω και το σαλιγκάρι της διαφάνειας και θέλουμε επενδύσεις, επενδυτικά σχέδια για την Ευρώπη, για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις επίσης και το ρυθμό των μεταρρυθμίσεων ακούσαμε από τον ΩΣΑ και τι μπορούμε να κάνουμε για να επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις και αναθέθηκε και εναρμόνιση και ενίσχυση της ενιαίας αγοράς. Ε, δεν αναφέρω όλες τις συστάσεις μίας προς μία, απλώς σας κάνω μια περίληψη. Τώρα λοιπόν έχετε το λόγο για να μας πείτε τις απόψεις σας και θα θέλαμε επίσης ε, να απαντάτε και ο ένας τον άλλον ε, αν θέλετε. Υπάρχει κάποιος ο οποίος θα ήθελε να ξεκινήσει, να κάνει την πρώτη δήλωση. Θα σας λέω με αριθμό, βλέπετε ποια θέση είστε, το 66 από το Route 66. Ε, έχετε το νούμερο στην οθόνη, μπορείτε να πατήσετε και το μικρόφωνο σας. Ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια για τις εξαιρετικές παρουσιάσεις και οι δύο ήταν ε, πάρα πολύ καλά διαρθρωμένες και θα ήθελα να προσθέσω ένα επιπλέον στοιχείο. Το στοιχείο αφορά τις επενδύσεις και επικεντρώνεται στις ιδιωτικές επενδύσεις. Όταν ε, λαμβάνεται απόφαση για επενδύσεις, το βασικό στοιχείο είναι το κόστος της χρηματοδότησης και μέσω της κρίσης αυτό το οποίο διαπιστώσαμε ήταν ότι για πολλές ε, περιφέρειες της Ευρώπης το κόστος της χρηματοδότησης ήταν υψηλότερο από το ε, ε, κεφάλαιο το οποίο επενδυόταν. Επομένως, η απόφαση να επενδύσει κάποιος αμφισβητείται όταν αντιστρέφεται η σχέση αυτή. Σε πολλές περιπτώσεις το κόστος της χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις είναι κάτω από το ε, κεφάλαιο το οποίο επιστρέφεται. Επομένω, αυτό αποτελεί επιπλέον κίνητρο. Και θεωρώ ότι αυτά τα δύο στοιχεία είναι πολύ σημαντικά όταν θέλουμε να δώσουμε όθηση στι επενδύσει. Δεύτερον, γνωρίζουμε επίση ότι το κόστο τη χρηματοδότηση δεν είναι ομοιόμορφο σε όλη την ένεση, που σημαίνει ότι ε, η δυνατότητα να διακρίνουμε το κόστος ε, χρηματοδότησης ε, ε, του πιστοτικού κινδύνου δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Και γιατί αυτό, διότι υπάρχει ακόμα επιμόλυνση από το κυρίαρχο κόστος χρηματοδότησης στην Ευρώπη για τον ε, τραπεζικό κίνδυνο και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλο, ε, μεγαλύτερο κόστος χρηματοδότησης για επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Νότια Ευρώπη. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να επιστρέψουμε λοιπόν σε εμείς τις επιχειρήσεις μας να μπορέσουν να αυξήσουν την δυνατότητα χρηματοδότησης τους ε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Ευχαριστώ. Θα ήθελε κάποιος να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Το 61. Συγγνώμη που σας λέω με τα νούμερα. Το 62 μάλλον. Έχετε κάποια απάντηση στο κόστος χρηματοδότησης. Όχι, είναι κάτι διαφορετικό. Υπάρχει κάποιος ο οποίος θα θέλει να απαντήσει στο θέμα του κόστου της χρηματοδότησης και πώς ε, μπορούμε να κάνουμε το κόστος κινδύνου σε κόστος κεφαλαίου. Βλέπω εδώ οι ομιλητρίες μας θέλουν να απαντήσουν. Το 62, παρακαλώ, ο κύριος και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστώ τις δύο κυρίες, κυρίες εισηγήτριες για όσα ακούσαμε και μας έδωσαν επαρκή χρήσιμα ε, στοιχεία προς αξιοποίηση. Η παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έφερε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη τη αντιμέτωπου με το πρόβλημα του ιδιαίτερα χαμηλού επίπεδου των επενδύσεων. Σε σύγκριση με το επίπεδο ρεκόρ του 2007, όπω αποδείχθηκε από τα στοιχεία των πινάκων, οι επενδύσει στην Ευρωζώνη μειώθηκαν κατά 15,6% κατά τη διάρκεια τη κρίση, ποσοστό το οποίο ανέρχεται σε 40-50% σε χώρε τη Νότια Ευρώπη. Οι ανεπαρκεί επενδύσει επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη με αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα να πλήττονται η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα των οικονομιών. Το κεφαλαιακό απόθεμα επηρεάζεται επίση σημαντικά συνιστώντα τροχοπέδι για το αναψιακό δυναμικό τη Ευρώπη και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασία. Στη χθεσινή τοποθέτησή του ο Πρόεδρος Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Γιούγκερ, αναφέρθηκε σε δύο βασικού πυλώνες, άξονε της λύσης του ελληνικού κορυφαίου οικονομικού προβλήματος, δηλαδή τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις. Ακούσαμε επίσης ε, ε, από την τοποθέτηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Σούλτς ε, την τοποθέτησή του για δραματική κρίση στην Ελλάδα λόγω των προσφύγων. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι η Επιτροπή έχει οθετήσει μια σειρά προγραμμάτων και μέτρων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων από τον προπολογισμό τη Ένωση. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μα τι τοποθετήσει αυτέ και τι επισημάνσει που έχουν γίνει, ώστε οι διαπιστώσει αυτέ να συμβάλλουν στι πρωτοβουλίε που θα αναλάβουμε για την επίλυση του προβλήματο. Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη ε, στοχεύει στην άρση των υφιστάμενων εμποδίων στι επενδύσει. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το σχέδιο Juncker, βρίσκεται στον πυρήνα αυτού του σχεδίου Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δίνεται σε αυτό σε έργα που αφορούν τομείς όπως η εκπαίδευση, η έρευνα, η καινοτομία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση και οι υποδομές. Απαιτείται μια ολοκληρωμένη και συλλογική προσέγγιση του προβλήματος των χαμηλών επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των αμεληταίων δυστυχώς σήμερα επενδύσεων σε χώρες όπως η Ελλάδα. Οφείλουμε να μεγιστοποιήσουμε τα ωφέλη της ενιαίας αγοράς οφείλουμε να είμαστε ευέλικτοι στην έγκριση κονδυλίων, παρακάμπτοντας τα γραφειοκρατικά εμπόδια και να μην εξαντλούμε την αυστηρότητά μας μέχρι τέλους. Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε με αποδοτικό και διαφανή τρόπο τα υφιστάμενα εμπόδια στον τομέα των επενδύσεων, στην ελεύθερη κίνηση των κεφαλαίων και στην προσέλκυση της συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών, ώστε να επανέλθουν οι ευρωπαϊκοί λαοί σε σταθερή τροχιά οικονομικής ανάκαμψη και ανθεκτικότητας με όπλο όλα τα προηγούμενα θα προχωρήσουμε στην παγκόσμια σκηνή με ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις όπως ελέγχθηκε λίγο πριν, συμμετέχοντας με εξωστρέφεια στο διεθνές εμπόριο και στις επενδύσεις. Και κλείνω λέγοντας ότι για να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί έναντι χωρών με χαμηλότερο κόστος παραγωγής χρειάζεται να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα. Μόνο έτσι... Μόνο έτσι θα δημιουργηθεί ένας ε, χώρος σταθερότητας και ευημερίας για όλους τους πολίτες της ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα για χώρες που αντιμετωπίζουν τελευταία τη μεγαλύτερη πρωτόγνωρη κρίση όπως είναι η Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Άκουσα μια σαφή δήλωση από εσά ότι το επενδυτικά σχέδιο, το, το σχέδιο στρατηγικών επενδύσεων ήταν ένα ουσιαστικό στοιχείο. Ε, θέλει κάποιος να απαντήσει σε αυτόν. Σαφώς εσείς είστε θετικά διακείμενος. Θα ήθελα να ακούσω περισσότερες απόψεις για το σχέδιο στρατηγικών επενδύσεων. Το 154. Μπορείτε να μας πείτε το όνομά σας και από ποιο κοινοβούλιο είστε από τη Γερμανική Βουλή. Συμφωνώ απόλυτα με τον Έλληνα Σνάλφο σε ένα θέμα. Χρειαζόμαστε περισσότερε ιδιωτικέ επενδύσει. Το σχέδιο Juncker και όλα τα μέτρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικά, αλλά δεν υποκαθιστούν τι ιδιωτικέ επενδύσει. Και οι ιδιωτικέ επενδύσει μπορούν να προκύψουν μόνο αν υπάρχει εμπιστοσύνη. Και η εμπιστοσύνη και η σταθερότητα. Αυτά χρειάζονται. Όταν έχω μια κυβέρνηση η οποία δρά με τρόπο αξιόπιστο, όταν έχω μια διοίκηση δημόσια που δρά με τρόπο αξιόπιστο. Όταν έχω εργαζόμενους που δεν κάνουν απεργία κάθε τρεις εβδομάδες. Όταν υπάρχει εμπιστοσύνη στον τρόπο παραγωγής και στη χώρα. Αυτό είναι το σημαντικότερο που πρέπει να κάνουμε, να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη στην Ευρώπη. Και μπορεί να δημιουργηθεί μόνο εάν θέλουμε από κοινού να αντιμετωπίζουμε τις κρίσεις. Κάτι άλλο που ανέφερε ο Έλληνας συνάδελφος. Είναι επίσης η μεταναστευτική κρίση που θίγει την Ελλάδα όπως και τη Γερμανία, την, την Σουηδία και, και άλλες χώρες. Αν θέλουμε λοιπόν ιδιωτικές επενδύσεις να υπάρξουν πρέπει να δημιουργήσουμε κλίμα εμπιστοσύνης. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να επιλύουμε από κοινού τις κρίσεις. Δεν θα λύσουμε την κρίση και δεν θα υπάρξουν επενδύσεις ούτε στην Ελλάδα, ούτε στις χώρες των Βαλκανίων, ούτε αλλού, εάν δεν λύσουμε το πρόβλημα της μετανάστευσης. Και γι' αυτό κάνω έκκληση να συνεχιστεί η κοινό συμφωνηθήσα εδώ στι Βρυξέλλε προσπάθεια μεταρρυθμίσεων, να είμαστε αξιόπιστοι και στη συνάντηση κορυφή αύριο και μεθαύριο να αντιμετωπίσουμε τα ε, προβλήματα που έχουμε ενώπιόν μα. Ωραία, σας ευχαριστώ. Επομένως, ε, εσείς δεν θέλετε απλώς ε, το στρατηγικό σχέδιο επενδύσεων να αντικαταστάσει τις ε, επενδύσεις, αλλά θέλετε εμπιστοσύνη. Αυτό άκουσα από την αγγλική μετάφραση 100 φορές. Χρειάζεται λοιπόν εμπιστοσύνη. Θέλει κάποιος άλλος να σχολιάσει το θέμα του επενδυτικού σχεδίου. Το 9. Πέστε μας το όνομά σας και από ποιο κοινοβούλιο είστε. Ντουρ από τη Γερουσία των Κατοχωρών συζητούμε την ανάγκη για ιδιωτικέ επενδύσει. Θα ήθελα να απαντήσω απευθείας στον Γερμανό συνάδελφο και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο χρειάζεται εμπιστοσύνη, είπε. Αλλά νομίζω ότι πρωτίστως οι επιχειρήσεις που έχουν αρκετά χρήματα για να επενδύσουν, εν γέννη, πρέπει να είναι βέβαιοι ότι θα υπάρχει ζήτηση για να πουλήσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θα παράξουν. Και το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να επενδύσουμε και τι είδους επενδύσεις χρειαζόμαστε προκειμένου να έχουμε ανάπτυξη που να περιλαμβάνει τους πάντες και θα διασφαλίζει και τη μελλοντική διζήτηση και θα είναι κατανεμημένη κατά τρόπον ώστε οι επενδυτές να μπορούν να βρουν καταναλωτές για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είδα και το 31 που θέλει να απαντήσει. Παρακαλώ το όνομά σας και από ποιο κοινοβούλιο έχετε. Από την Εσθονία. Συμφωνώ με του συναδέλφου για τι ιδιωτικέ επενδύσει. Αυτέ δημιουργούν ανάπτυξη στην ουσία. Και αν συζητήσει κανεί με έναν επιχειρηματία, ε, αναφέρονται πάντα στην έλλειψη εμπιστοσύνη και υπάρχει ένα ερωτηματικό. Τι θα συμβεί. Αυτό σχετίζεται με ε, τις επιχειρήσεις και το συνολικό παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, μεν, αλλά πρόσφατα αυτό το οποίο διαπιστώσαμε είναι ότι έχει σχέση και με την πολιτική κατάσταση. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην ε, μεταναστευτική κρίση, αλλά και τα όσα συνέβησαν στη Ρωσία και συμβαίνουν ακόμα. Θεωρώ λοιπόν ότι ε, πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα ώστε να μειώσουμε αυτούς τους κινδύνους. Το δεύτερο είναι ότι είναι πιο εύκολο στην ουσία να λάβει κάποιος δανειοδότηση οι ιδιωτικά κονδύλια για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Το πρόβλημα είναι για τις μικρότερες επιχειρήσεις και οι μικρές επιχειρήσεις στην Εστονία είναι πολύ μικρές σε ευρωπαϊκούς όρους. Με 20 υπαλλήλους ε, έχει κάποιο μία μεσαία επιχείρηση. Ε, περί αυτού πρόκειται. Επομένω, για αυτού είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρουν χρηματοδότηση, ακόμα και αν είναι χαμηλά τα επιτόκια. Γιατί οι τράπεζε, που είναι διεθνεί τράπεζε, ακόμα ανησυχούν για πάρα πολλά ζητήματα τα οποία δεν σχετίζονται με την ίδια την Εστονία αλλά με όλη την Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε και αυτούς τους κινδύνους. Και από τις παρουσιάσεις που ακούσαμε εγώ ως οικονομολόγος θα ήθελα να συζητήσω πολλά από τα θέματα που θίξατε εσείς στις παρουσιάσεις αλλά δεν έχουμε χρόνο βεβαίως. Εξακολουθώ όμως να πιστεύω ότι αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα εξετάσουμε και να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε όλους αυτούς τους κινδύνους ε, που υπάρχουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σαφές λοιπόν ότι μας ενδιαφέρει η εμπιστοσύνη να επιλύονται τα προβλήματα από κοινού, όχι μόνο τα γεωπολιτικά αλλά και τα οικονομικά προβλήματα. Ε, Θέξατε και το θέμα της χρηματοδότησης, τον οποίο έθιξε και η κυρία Φανχέστ, ε, κυρίως για την ε, ε, χρηματοδότηση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχει κάποιος ο οποίος θα ήθελε να σχολιάσει κάτι από αυτού, να κάνει μια σύσταση, μια δήλωση, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ρούμαν Γκέτσιφ από το Κοινοβούλιο της Βουλγαρίας δύο πράγματα. Πρώτον, οι ιδιωτικέ επενδύσεις και οι δημόσιες επενδύσεις ε, είναι εντελώς διαφορετικές υποθέσεις. Αν ε, τα εξετάσετε αυτά ως ε, δυνατότητα ΣΔΙΤ, σύμπραξης δημοσίου ιδιωτικού τομέα, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Οι δημόσιες επενδύσεις υπολογίζεται τρει ή τέσσερι φορέ εάν υπάρχει δυνατότητα από τη δημόσια επένδυση να προσελκύσει ιδιωτικέ επενδύσει. Επομένω, ε, μεγάλε επενδύσει, ακόμα και στη βιομηχανία, που θα ξεκινήσουν με κίνητρο το σχέδιο ε, Juncker, σίγουρα θα βοηθήσουν ε, θετικά στην οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Επίσης θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις ε, λεγόμενες τράπεζες που θα πρέπει να ενθαρρύνουν, διότι όλοι αναφέρονται στις ιδιωτικές επενδύσεις και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν δυσκολία πρόσβαση στην ε, ε, χρηματοδότηση και επομένως θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια και οι κυβερνήσεις πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις τράπεζες που θα βοηθήσουν αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τι είδους τράπεζες είναι αυτές, πώς τις είπατε, αλλά κυρίως για τις μικρές εξειδικευμένες δημόσιες τράπεζες οι οποίες χρηματοδοτούνται από την ιδιωτική αγορά αλλά ε, δανειοδοτούν υπό πολύ συγκεκριμένες συνθήκες ε, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ. Καλή η πρότασή σας. Το 36 Πείτε μα όνομα και κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Φρανσέσκο Καριέλο, από το Ιταλικό Κοινοβούλιο. Θα τα πω Ιταλικά, συγγνώμη. Νομίζω ότι οι Ιταλικές επιχειρήσεις, προκειμένου να επενδύσουν, χρειάζονται λιγότερη γραφειοκρατία, πραγματικά επιτόκια τα οποία θα είναι βάση του πραγματικού πληθωρισμού στη χώρα στην οποία δραστηριοποιούνται και ασφάλεια. Αυτά απαιτούν οι ιδιωτικέ επενδύσεις και κατά την άποψή μα, το σχέδιο Juncker, το πιο μεγάλο σχέδιο επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επιτρέπει να συμβούν όλα αυτά. Το σχέδιο ε, θα έπρεπε να προσελκύει ιδιωτικέ επενδύσεις, αλλά κατά την άποψή μα θα έπρεπε να, να αποφύγει, συγγνώμη, να δημιουργήσει δεσπόζουσε θέσει στην αγορά και να υπονομεύσει τον ανταγωνισμό διότι επενδύοντας σε ιδιωτικές επενδύσεις, επομένως διευκολύνοντας κάποιες επιχειρήσεις να επενδύσουν σε ιδιωτικές υποδομές, δημιουργούνται και συνθήκες ε, κρατικής επιχορήγησης προς κάποιους ε, ε, φορείς του ιδιωτικού τομέα, αντί να διευκολύνουμε τον ανταγωνισμό. Ταυτόχρονα, κάποιες άλλες επιχειρήσεις θα μπορούσαν την ίδια παρέμβαση ε, να υπονομεύονται ως προς τη δυνατότητά τους να επενδύσουν στην ίδια δομή. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν επενδύσεις ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία και να διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται με πλήρη ανταγωνισμό και επίσης όρι σε όλα τα επίπεδα. Your feelings about Ωραία, εσείς είστε λιγότερο ζεστός συνεπώς από ότι οι υπόλοιποι, να το συνοψίσω έτσι. 383. Εσείς παρακαλώ. Ευχαριστώ. Βλέπα. Σφίκλα από την Σλοβενία. Και πολύ χαίρομαι γιατί εδώ δεν τίθεται το ερώτημα ναι ή όχι στις επενδύσεις. Η απάντηση είναι σαφής. Προφανώς και χρειαζόμαστε επενδύσεις. Φυσικά και θα ήθελα και εγώ επενδύσει σε όλους τους τομείς υποδομών. Χρειαζόμαστε κτίρια, διαμερίσματα, δρόμους, σειροδρομικές υποδομές κλπ. Γιατί έτσι ε, διευκολύνεται η μετακίνηση. Χαίρομαι λοιπόν για την ιδέα επίσης που είναι επένδυση στην εκπαίδευση. Γιατί όντω η προστιθέμενη αξία εδώ είναι τεράστια κυρίως για την αγορά εργασία στη συνέχεια. Όμως πρέπει να αναρωτηθούμε μερικά πράγματα και να δώσουμε και απαντήσεις βέβαια. Γιατί χρειαζόμαστε επενδύσεις. Χρειαζόμαστε επενδύσεις επειδή έχουμε χρεωθεί τόσο πολύ και πρέπει να μειωθεί το χρέος μας. Και είναι προϋπόθεση για μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη. Επίσης, η απασχόληση και η κοινωνική πολιτική. Είναι πολύ σημαντικό εδώ να διασφαλίσουμε ότι τα επίπεδα απασχόλησης θα αυξηθούν και θα μειωθεί η ανεργία συνεπώς. Άρα ερχόμαστε στο άλλο. Ποιος πρέπει να επενδύσει. Ο δημόσιος τομέας και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να επενδύσουν. Η αναλογία θα πρέπει να είναι σωστή φυσικά. Όμως δεν είναι ξεκάθαρο για μένα πόσο θετικό είναι το θέμα της εταιρικής σχέσης δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Πανέρχομαι στο ότι επενδύσει τις χρειαζόμαστε παντού, πάντα, αλλά πώς, πώς να επενδύσουμε. Εδώ τίθεται δύο ερωτήματα. Πρώτον, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές όσον αφορά τις προσδοκίες μας από τις επενδύσεις. Δεν μπορεί να περιμένουμε αύριο ή μεθαύριο να αποδώσουν οι επενδύσεις μας. Μερικές επενδύσεις χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να αποδώσουν. Δεύτερον, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το κράτος και οι τράπεζες να διευκολύνουν τις επενδύσεις. Ο τραπεζικός τομέας είναι υπεύθυνο για την κρίση του 2008, οπότε θα έπρεπε να δραστηριοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Θα έπρεπε οι τράπεζες να διευκολύνουν τους επενδυτές Πώς προσφέροντας ε, βέβαια χαμηλά επιτόκια. Και όσον αφορά το κράτος, το κράτος από τη δικιά του την πλευρά πρέπει να διασφαλίσει ότι κάποιοι φόροι, τέλη μειώνονται για τους επενδυτές. Πρέπει βέβαια να μειωθεί και η γραφειοκρατία όσο γίνεται περισσότερο. Εννοείται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Τελευταίος εδώ μπροστά. Ο κύριος 2.83, εσείς. Και μετά θα ζητήσουμε απαντήσει από το πάνελ. Εγώ Πίμινεφ, από την Λετωνία, τη ΣΑΙΜΑ, το Εθνικό Κοινοβούλιο της Λετωνίας. Συζητάμε εδώ για τράπεζες, οι οποίες θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν από το κράτος. Δεν είναι τράπεζες που ανήκουν στο κράτος τελικά και που δεν απαγορεύεται αυτό από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Τα δημόσια κονδύλια άρα πρέπει να επενδυθούν στο κεφάλαιο ε, της τράπεζας, οπότε η τράπεζα να μπορέσει να βρει και άλλα χρήματα και έτσι να υπάρξει κίνηση στην εθνική αγορά με τη μορφή δανείων. Δεν θα υπάρχει καθόλου πληθωρισμός. Τα δάνεια θα δίνονται στα πλαίσια των προγραμμάτων ανάπτυξης και όχι για δαπάνες. Δεν... Ε, είναι πολύ σημαντικό για χώρες όπως είναι η Λετωνία, για παράδειγμα, από όπου έρχομαι εγώ. Αυτό θα συνεισφέρει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητα της χώρας. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι η κατάσταση στη δικιά μου τη χώρα, τη Λετωνία, θυμίζει πολύ την κατάσταση στη Γερμανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Γερμανοί επιχειρηματίες δεν είχαν χρήματα, δεν είχαν ασφάλεια και λίγοι δούλευαν. η Γερμανία έλυσε αυτή την κατάσταση δημιουργώντας ε, κρατικές τράπεζες ή τράπεζες που ανήκαν στις τοπικές ε, κυβερνήσεις. Για τις χώρες λοιπόν αυτές που βγαίνουν από την κρίση, μια τέτοια ανάπτυξη με κρατικές τράπεζες είναι μια καλή λύση γιατί έτσι ρίχνονται επενδύσεις στην οικονομία. Ωραία. Απαντήσεις από το πάνελ τώρα. Ακούσαμε πολλές παρατηρήσεις για τις επενδύσεις, για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, την πρόταση για κρατικές επενδυτικές τράπεζες, χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παρακαλώ, κύριε Κιβινιέμι. Ευχαριστώ για τα πολύ ενδιαφέροντα σχόλια της ζωντανή συζήτηση και ε, πολύ χρήσιμα τα θέματα που αναφέρατε. Για το θέμα της εμπιστοσύνης. Όντως, η έλλειψη επενδύσεων οφείλεται στην έλλειψη εμπιστοσύνης. Και έχουμε κάνει και εμείς διάφορες μελέτες που το αποδεικνύουν. Οι εταιρείε ε, διστάζουν να επενδύσουν. Είναι οι αβεβαιότητες που υπάρχουν για το τι πολιτική θα υπάρξει και τι ρυθμιστικές διατάξεις. Πρέπει λοιπόν να το αντιμετωπίσετε για να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις που έχετε μπροστά σας, όπως για παράδειγμα το προσφυγικό. Ε, παρακαλώ μην επιτρέψετε να καταρρεύσει το Σέγγεν. Δεν θα ήταν καλό. Αλλά αν κοιτάξουμε με ένα στοιχεία από τα τελευταία χρόνια, θα μπορούσαμε να έχουμε μεγάλες δυσχέρειες να καταλάβουμε γιατί είναι τα στοιχεία έτσι. Δηλαδή, τα επιτόκια είναι πολύ χαμηλά. Η ισοτιμία του ευρώ πέφτει και η τιμή του πετρελαίου πέφτει. Πέρυσι λοιπόν, για αυτούς τους λόγους, η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη θα έπρεπε να ήταν κατά 1% μεγαλύτερη και όμως δεν ήταν. Και αν δούμε την τελευταία πεντηκονταετία μόνο για μια πενταετία η ανάπτυξη του εμπορίου ήταν χαμηλότερη από την ανάπτυξη του ΑΕΠ ενώ τα περισσότερα άλλα χρόνια ήταν μεγαλύτερη. Πέρυσι όμως δεν είχαμε ύφεση ενώ σε όλες τις άλλες περιόδους που η ανάπτυξη του εμπορίου ήταν μικρότερη από την ανάπτυξη του ΑΕΠ, είχαμε ύφεση. Καταλαβαίνω αυτούς που λένε ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις ε, θέλουν να μην υπάρχει αβεβαιότητα. Ξέρετε πέρυσι, ακόμη και στις Ηνωμένε Πολιτείε οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να έχουν επενδύσει διπλάσια ποσά αν δούμε τι ποσά είχαν ως αποθέματα στις τράπεζες χωρίς δηλαδή να χρειαστεί να πάρουν δάνειο ίδια λοιπόν είναι η εικόνα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη τι θα μπορούσε να κάνει λοιπόν ε, η Ένωση θα μπορούσε να εμβαθυνθεί η ενιαία αγορά και να βελτιωθεί η λειτουργία της εξετάσαμε από μια οπτική γωνία την ενιαία αγορά από τον τομέα των υπηρεσιών. Χρειάζεται πιο φιλόδοξη εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Μόνο αυτή θα μπορούσε να προκαλέσει μία αύξηση της τάξης του 0,6 έως 2% του ΑΕΠ μακροπρόθεσμα. Και αυτό είναι μόνο ένα τμήμα τη οικονομίας. Καλύτερη λειτουργία λοιπόν της ενιαίας αγοράς, εμβάθυνσή τη. Αυτά χρειάζονται. Αναφερθήκατε στην Ενεργική Ένωση, την Ένωση Κεφαλαίων Αγορών και την ψηφιακή ενιαία αγορά. Και αυτά θα βοηθούσαν. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο. Ωραία, θα επανέλθουμε στην εμβάθυνση της ενιαία αγορά. Αφού πρώτα ακούσουμε την κυρία Χέστ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σα. Συμφωνώ με τον Ωσα ότι η εμπιστοσύνη είναι θεμελιώδε. Όμως έχουν υπάρξει διαφορές ε, εντός τη Ένωση. Ορισμένες χώρε έχουν κάνει περισσότερα βήματα για να επανέλθει η εμπιστοσύνη. Άρα δεν είναι συνολικά μελανή η εικόνα. Αν κάνει αυτό που πρέπει, αμείβεσαι για να βγάλουμε και κάτι θετικό. Όμως δεν υπάρχει μαγική συνταγή. για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει ζήτηση, είτε στη χώρα σας είτε στο εξωτερικό δυνατότητες διάθεσης και επίσης οι επενδύσεις τους να μην αντιμετωπίζουν ε, γραφειοκρατικά εμπόδια και δυνατότητες δανειοδότησης. Ας συγκρίνουμε την Ένωση με τις Ηνωμένε Πολιτείες, πώς επέλυσαν την ε, τραπεζική κρίση με πολύ διαφορετικό τρόπο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρξε σχετικά σύντομη εξυγίανση, ενώ εμείς ε, καθυστερούμε. Και επειδή χρειάζεται ακόμη εξυγίανση αρκετών τραπεζών, θέλω να σας παροτρύνω να μην καθυστερήσετε περαιτέρω. Κάντε γρήγορα. Όσο πιο γρήγορα τις εξηγιάνεται, τόσο πιο γρήγορα θα αρχίσουν να δανειοδοτούν την οικονομία. Και ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Τέτοιο πρόβλημα έχουμε και στην Ολλανδία. Και δεν είναι εύκολο να το επιλύσει κανείς Οι μικρομεσαίες ε, εν γενός είναι πιο επικίνδυνες Άρα είναι πιο δύσκολο να δανειοδοτηθούν. Λαμβάνουν ε, μικρότερες επίση δανειοδοτήσεις άρα το διοικητικό κόστος είναι μεγαλύτερο αναλογικά. νομίζω ότι κατά ανάγκη ο σωστό τρόπος είναι να υπάρχουν κρατικές τράπεζες. Πρέπει να αποδείξουμε ότι θα είναι πιο αποτελεσματικές. Ο καθένας θέλει να επενδύσει εκεί που θα έχει την καλύτερη απόδοση. Οπότε, ναι μεν οι κρατικές τράπεζες επενδύσεων μπορούν να λειτουργούν με διάφορους τρόπους, αλλά πρέπει να αποφύγουμε οι κρατικές τράπεζες και δεν θέλω να, προσβάλλω κανένα από τους παρευρισκόμενους οι κρατικές τράπεζες δεν θα επενδύουν ε, σε πολιτικά σκόπιμα αλλά σε οικονομικά σκόπιμα ε, επενδυτικά προγράμματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για αυτή την τελευταία παρατήρησή σας για τις ε, επιχειρήσεις. Νομίζω ότι αυτό συνάδει με τις παρατηρήσεις που έγιναν εδώ και στην ε, ε, πρώτη σειρά οι ε, κρατικές τράπεζες ε, δεν βοηθούν για το ιδιωτικό κεφάλαιο. Άλλες παρατηρήσεις εδώ μπροστά το όνομά σας και από ποιο κοινοβούλιο είστε. Γιώρης Μπάχεμ από την Ολλανδική Γερουσία. Όσο περισσότερο ακούω την ομιλήτρια από τον ΩΣΑ, αυτό το οποίο με εντυπωσιάζει είναι ότι ευθύς εξ αρχής η ενιαία αγορά και η ολοκλήρωση ήταν κάτι που ήταν στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν εξετάσει κανείς τις επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις αναζητούν κλίμακα, ελεύθερη αγορά. Και υπάρχουν κάποιες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που με κανένα τρόπο δεν θα καταφέρουν να προσελκύσουν αυτές τις επενδύσεις. Θα προσελκύσουν επενδύσεις ε, στις μεγαλύτερες περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα γίνει εάν οι αγορές είναι πιο εναρμονισμένες. Έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε διάδοση και να υπάρχει όφελος για όλους πιο ουσιαστικά και πιο σωστά. Η εναρμόνιση είναι λοιπόν στο επίκεντρο αυτών που πρέπει να συμβούν και αν δω και το σχέδιο Juncker νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ε, ισχυρή όθεση, ένα σχέδιο Juncker Sin για να μπορέσουμε να πάμε σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε στην πραγματικότητα, δηλαδή μια νέα αγορά. Η διαδικασία αυτή από το 2005 και μετά καθυστερεί και δεν το συζητάει κανείς αυτός και χαίρομαι που το θίξατε γιατί αυτό είναι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό γιατί και η κυρία Κιβινιέμι ήταν απόλυτα σαφής ε, σε όλους μας και στους ε, βουλευτές και στους ευρωβουλευτές ότι ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων και της εναρμόνισης μειώνεται. Επομένως υπάρχει σαφής ανάγκη για δράση και επιτάχυνση από ό,τι άκουσα και από τις δύο μιλήτριες. Θέλω να προσθέσω και το εξή. Νομίζω ότι η δομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής που ε, επικρίνεται πολύ είναι όμως αυτοί οι οποίοι είναι ικανοί να εναρμονίσουν την οδηγία για τις υπηρεσίε και άλλους τομείς και δεν βλέπω να γίνεται κάτι παρά το γεγονό ότι τα ηχέγγυα υπάρχουν. Ίσως όχι η πολιτική βούληση. Αυτό ίσως θα έπρεπε να ενθαρρύνουμε. Άλλος κανεί για την επιτάχυνση της εναρμόνισης και τη εμβάθυνση τη εσωτερική αγορά. Απόψεις επ' αυτού. Κάποια άλλη πρόταση. 149 ο κύριος, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Από την Γερουσία της Τσεκιεχίας. Θα ήθελα να ξαναπάμε λίγο στο Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και αυτή της μορφής ε, της επενδυτικής επενδυτικές η γερουσία μα ε, θεωρεί ότι είναι θετικό εργαλείο για να πολλαπλασιάσουμε τις ιδιωτικές επενδύσεις ε, ε, και τις δημόσιες επενδύσεις με ιδιωτικά μέσα. Εμείς στην περιοχή μας έχουμε βιομηχανικέ περιοχές και αυτό αποτελεί κίνητρο για τους ξένους επενδυτές, αλλά δεν αρκεί. Στην Ευρώπη των 28 να πηγαίνουμε ένα στη βιομηχανική περιοχή του άλλου και να επενδύουμε. Ε, έχουμε καλέσει για παράδειγμα την Κορέα. Έχουμε τώρα Κινέζους επενδυτές. Παράγουμε το ε, Ιώτα, Citroën, Peugeot, αυτοκίνητα αυτών των τριών ε, βιομηχανιών και το καθεξής. και αυτό το οποίο θα θέλαμε για το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων είναι, μιας και λέμε για τις επιθυμίες μας, είναι να υπάρχει ένα κριτήριο διαφάνειας για τα επιλέξιμα έργα. Έργα τα οποία θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει επίσης να είναι το σωστό κριτήριο η διαφάνεια όταν ε, γίνεται η επιλογή των έργων. Ε, αυτό το οποίο πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη είναι κατά πόσον μπορεί να συνδυαστεί με άλλα θεματικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα τον ορίζοντα 2020. Εμείς είμαστε μικρή χώρα, αλλά θεωρούμε ότι αυτό είναι το λογικό έχουμε συντάξει και μια επιστολή την οποία θα διαβάσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υποστηρίζουμε το πλαίσιο του ε, Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων για το 2018. Ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει στην ανάπτυξη, στην απασχόληση και στην ευρωπαϊκή οικονομία. Άρα, μας ξαναφέρνετε στο Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το οποίο υποστηρίζεται Σαφέστατα, ε, για το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ή για κάτι άλλο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, το όνομά σας και από ποιο κοινοβούλιο είστε. Από το Φιλανδικό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Εξαιρετικές οι παρουσιάσεις που ακούσαμε σήμερα από τις ομιλήτριες. Πράγματι, οι επενδύσεις ε, είναι ουσιαστικής ε, για την ανάκαμψη και τις θέσεις εργασίας στην Ευρώπη ε, και την ανάπτυξη και ε, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει απαραίτητη εμπιστοσύνη για να ξεκινήσει η ροή των επενδύσεων. Χρειαζόμαστε ότι πρέπει να, θεωρούμε συγγνώμη, ότι πρέπει να υπάρχουν επενδύσεις καθαρής ενέργειας και έχουμε ξεκινήσει ήδη. Ποια είναι η άποψή σας επ' αυτού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επενδύσει ε, λαμβάνοντας υπόψη και την κλιματική αλλαγή, τις ε, βιοοικονομίες και τις καθαρές ε, επενδύσεις ενέργειες. Ωραία, να την αφήσουμε στην άκρη λίγο αυτή την ερώτηση προς το παρόν. Το ερώτημα είναι κατά πόσον τα επενδυτικά προγράμματα θα πρέπει να είναι για ε, καθαρές τεχνολογίες. Θα επανέλθουμε στο πάνελ μας μετά την επόμενη ερώτηση από τον κύριο στο 347. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι από το Ουγγρικό Κοινοβούλιο και θα ήθελα να σας πω για τη σωστή αναλογία ε, δανειοδοτήσεων και επιδοτήσεων. Εμείς θεωρούμε ότι η κατάλληλη ευρωπαϊκή προσέγγιση για την όθηση των επενδύσεων θα πρέπει να είναι ένα κατάλληλο μείγμα επιδοτήσεων και δανειοδοτήσεων, διότι επιδοτήσεις θα βοηθήσουν τις ε, λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες να ε, επιταχύνουν και να προσεγγίσουν τη συνοχή. Εμείς είμαστε υπέρ του προγράμματος οικονομικής ανάκαμψης που ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2014 και ε, χαιρετίζουμε και τους ε, στόχους επενδύσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να παραμείνουν και επιδοτήσεις όμως πέραν ε, των δανειοδοτήσεων, διότι υπάρχουν διαφορές ε, στο επίπεδο ανάπτυξης ε, των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προκειμένου να διασφαλίσουμε τη συνοχή χρειαζόμαστε και επιδοτήσεις. Ε, καλωσορίζουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων και θα θέλαμε να το χρησιμοποιήσουμε ως επιπλέον μέσο χρηματοδότησης. Πολλοί είπαν και εμεί συμφωνούμε ότι η διαδικασία χρηματοδότηση και η διαδικασία υποβολή αίτησης θα πρέπει να απλουστευτούν. Και πάλι παρατηρήθηκε για το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Να δώσουμε το λόγο στου ομιλήτριέ μας για να απαντήσουν. Όμως έγιναν και ορισμένε παρατηρήσεις για την ε, διαφάνεια και τα κριτήρια που θα εφαρμόσει το ΕΦΣΥ, το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Και άλλη ερώτηση. Το ΕΦΣΥ θα έπρεπε να επενδύσει σε επιχειρήσεις καθαρής τεχνολογίας. Η κυρία Κιβινιέμι. Ευχαριστώ. Όταν, ε, εάν θέλουμε να μιλήσουμε για τα πλεονεκτήματα της βιοοικονομίας, της κυκλικής οικονομίας, της οικονομίας ε, καθαρών τεχνολογιών μετά και την συμφωνία στο Παρίσι πριν από δύο μήνες, Όλα αυτά είναι μεγάλες προκλήσεις ε, συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να επιτύχει τους συμφωνηθέντες στόχους. Δεν θα το επιτύχει μόνη της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να συμβάλλουν και να επιτύχουν τους στόχους τους όλες οι χώρες του κόσμου. Σίγουρα υπάρχει πολύ δυναμικό εδώ, μεγάλες δυνατότητες και η Κομισιόν για την βιοοικονομία και την κυκλική οικονομία. Η Κομισιόν λοιπόν έχει παίξει μεγάλο ρόλο και προσπαθεί, να ενθαρρύνει και τα κράτη-μέλη. για να ευνοηθεί, να ανθίσει η βιοοικονομία και η κυκλική οικονομία. Είναι σίγουρα μία από τις λύσεις μέλλοντος. Τώρα για το ΕΦΣΙ δεν θα αναφερθώ στις λεπτομέρειες, γιατί αυτά είναι θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, επιδοτήσεις, ε, δανειοδοτήσεις, ε, διαφορετικές δυνατότητες. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω, ότι το ΕΦΣΙ θα πρέπει πραγματικά να σημαίνει προστιθέμενη αξία. Άρα επενδύσεις που να είναι κάπως υψηλότερου κινδύνου από τις προηγούμενες επενδύσεις που έχει χρηματοδοτήσει για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Να είναι κάτι καινούριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι όντως μια προσπάθεια που αξίζει. Και έτσι θα προσελκύσει και ιδιώτες επενδυτές. Με αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να λειτουργήσει. Και να αναφερθώ και σε κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε, Πρόεδρε. οικονομία χωρίς αποκλεισμούς. Ο ΩΣΑ έχει ασχοληθεί πολύ με αυτό το θέμα, οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Τι σημαίνει αυτό. Λέμε ότι πρέπει να υπάρξει απελευθέρωση στην αγορά και στην αγορά εργασίας, αλλά παράλληλα λέμε ότι χρειάζονται και συνοδευτικές πολιτικές. Δηλαδή πρέπει να μας απασχολήσουν και εκείνοι που λόγω αυτής της φιλελευθεροποίησης θα χάσουν τη δουλειά τους. Κάποιες επιχειρήσεις θα χρεοκοπήσουν. Θα πρέπει να δοθούν δυνατότητες επαγγελματικής κατάρτισης και άλλα συνοδευτικά υποστηρικτικά μέτρα για να βρουν και αυτή τη θέση τους κάπου αλλού στην αγορά εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό να ασχοληθούμε και με το επίπεδο κατάρτισης και τις δυνατότητες επαγγελματικής εκπαίδευσης και συνολικότερα με ένα πιο καινοτόμο σύστημα να έχουμε μια συνολική λύση για να μην υπάρξουν αποκλεισμοί. Ευχαριστώ κυρία Φανχέριστ. Σύμφωνα απόλυτα με αυτά που λέει συνάδελφος του ΩΣΑ. Αλλά και τα εξής θέλω να τονίσω. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο θέμα επενδύσεων. Είναι θέμα συνολικότερο περιβαλλοντικής πολιτικής. Το σύστημα εμπορίας εκπομπών, για παράδειγμα ρήπων, δεν λειτουργεί τόσο καλά. Άρα πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματικό. Στην Ολλανδία, αν κάνει κανείς μελέτη κινδύνου απόδοσης για αυτές τις επενδύσεις, δεν βγαίνει πολύ θετικό το αποτέλεσμα γιατί ο τρόπος που λειτουργεί το σχήμα εμπορίας ε, ρήπων δεν λειτουργεί. Στην Ολλανδία κάνουμε μια συζήτηση, βέβαια αλλού γίνεται περισσότερη συζήτηση, για την αύξηση των ανισοτήτων. Θεωρούμε ότι οι ανισότητες ε, αυξάνονται διότι ε, υπάρχουν λιγότερο υψηλού επίπεδου εκπαίδευση ε, άνθρωποι από ό,τι ανάγκες. Άρα, ε, μέσω επενδύσεων στην εκπαίδευση θα έχουμε διπλό θετικό αποτέλεσμα. Θα μειώσουμε τις ανισότητες. Ευχαριστούμε. Και δύο. Ανοίξατε τώρα τη συζήτηση προκειμένου να κοιτάξουμε πιο μακριά από τις επενδύσεις. Είπατε επίσης ότι πρέπει να επιταχυνθεί η δουλειά που γίνεται για τις μεταρρυθμίσεις. Αναφερθήκαμε και το σύστημα εμπορίας ρήπων. Θα ήθελα τώρα να δώσουμε το λόγο σε όσους εκπροσώπους εδώ θα ήθελα να σχολιάσουν πέρα από τις επενδύσεις, πέρα από το επενδυτικό ε, ταμείο στρατηγικών επενδύσεων. Τι άλλο. Εκτός από τις επενδύσεις πάνω στις οποίες σίγουρα πρέπει να δουλέψουμε πολύ, υπάρχουν λοιπόν και τα άλλα. Εσείς παρακαλώ. Εδώ μπροστά. Θέλω να ρωτήσω για τις δημόσιες επενδύσεις στην κυρία Κιβινιέμη. Δώσατε ένα επιχείρημα υπέρ περισσότερων δημοσίων επενδύσεων, ενώ η ομόλογό σας η Ολλανδές, είναι πιο επιφυλακτική. Στην Ολλανδία χρειάζεται μια ελάχιστη απόδοση 4,5% για τις δημόσιες επενδύσεις. Και αυτό οφείλεται στο πρίμιο του 3% και επειδή από πλευρά των φορολογούμενων ε, πολλά τελικά σχέδια δεν είναι αποδοτικά. Συμφωνείτε να υπάρχει αυτό το 3% risk premium, πριν κινδύνου. Και πώς αυτό συνδυάζεται με την άποψή σας ότι χρειάζονται περισσότερες δημόσιες επενδύσεις για να ενισχυθεί η οικονομική ανάπτυξη. Πρόεδρε, όταν μιλάμε για βραχυπρόθεσμα ε, μέτρα, πολλές ευρωπαϊκές χώρες και ακόμα και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια τέτοια εφαρμογή θα ενίσχυε την ανάπτυξη, την οικονομική, άρα χρειάζονται επενδύσεις. Υπογράμμισε όμως χρόνο ότι δεν θα πρέπει να είναι οτιδήποτε επενδύσει, πρέπει να τις εξετάζουμε, να είμαστε σίγουροι ότι η οικονομία μπορεί να αποφεληθεί από αυτές και ότι μακροπρόθεσμα αποδίδουν. Τα κριτήρια λοιπόν πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένα, να βάζουμε ψηλά τον πύχη. Η απόδοση μπορεί να είναι μετά από μερικά, μερικούς μήνες. Τα κριτήρια δεν θα πρέπει να είναι χαλαρά. Το ίδιο ισχύει και για τις μεταρρυθμίσεις. Το κύριο μήνυμά μου δεν είναι αυτό. Το κύριο μήνυμά μου είναι ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι αναγκαίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να μαθαίνουμε περισσότερο στην ενιαία αγορά. Και να επιταχύνουμε, ναι, αυτό είναι το μήνυμά σας. Άλλος. Ποιος θα ήθελε να σχολιάσει, να παρέμβει. Α, εσείς. 41. Παρακαλώ. Κερτελίνα, Αυστρία. Οι επενδύσεις είναι πολύ σημαντικές, αλλά το πιο σημαντικό είναι να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη. Και γι' αυτό χρειάζονται και ιδιωτικές και δημόσιες. Αλλά οι ιδιωτικές επενδύσεις δεν θα υπάρχουν εάν δεν βλέπουν να υπάρχουν δυνατότητε διάθεσης των προϊόντων τους. Δηλαδή, πολλές τράπεζες θα θέλουν να δώσουν περισσότερε περισσότερες ε, ε, χρηματοδοτήσει, αλλά οι επιχειρήσεις δεν βλέπουν να υπάρχει αγοραστική δύναμη. Η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών λοιπόν είναι εξίσου αναγκαία για αυτή την πολιτική για να προωθηθούν οι επενδύσεις και θα πρέπει η επιχείρηση να μπορεί να πουλήσει περισσότερα προϊόντα και να μπορεί να κάνει περισσότερες εξαγωγές. Τότε θα κάνω επένδυση ως επιχειρηματίας. Οι δημόσιες επενδύσεις. Συγχαίρω τον συνάλφα από τη Λετωνία ο οποίος πρότεινε να υπάρχει μια ιδιωτική τράπεζα επενδύσεων. Αλλά το θεμελιώδες ερώτημα είναι πού θα βρούμε τα λεφτά. Γιατί πρέπει πάντα η αναχρηματοδότηση να γίνεται μέσω ιδιωτικών τράπεζων, τραπεζών. Θα το καταλάβαινα. Εάν οι τράπεζες θα ήθελαν να διαθέσουν για δημόσια ε, προγράμματα τα χρήματα των φορολογουμένων. Αλλά στην ουσία δεν το κάνουν. Γιατί όμως εφόσον οι ιδιωτικές τράπεζες δεν το κάνουν δεν δημιουργούμε μια δημόσια τράπεζα για να το κάνει. Διότι αν μια τράπεζα θέλει, μια δημόσια τράπεζα θέλει να, να χρηματοδοτήσει το χρέος της τότε μπορεί να βγάλει ομόλογα και τα ομόλογα βασίζονται τα κρατικά εισοδήματα και τα κρατικά εισοδήματα βασίζονται στην εργασία των πολιτών. Μπορεί λοιπόν μια δημόσια τράπεζα να χρηματοδοτήσει τις επιχειρήσεις και μετά τα μερίσματα, τα κέρδη που θα βγάλει μια δημόσια τράπεζα θα είναι δημόσια έσοδα. Θα είναι προς όφελος των πολιτών. Προς όφελος των πολιτών. Και μπορεί να δημιουργήσει κεφάλαιο μια δημόσια τράπεζα. Θα μπορούσαν για παράδειγμα να εκδοθούν ε, ομόλογα που να συνδέονται με το ΑΕΠ που να βασίζονται και να συνδέονται με την ανάπτυξη, με τα ποσοστά ανάπτυξης. Δεν ξέρω αν ε, το ρώτησε, το έθεσε έτσι ο συνάδελφος, αν μπορούμε μέσω σύνδεση με το ΑΕΠ να χρηματοδοτήσουμε. Ναι, όντω υπήρχε αυτή η στήριξη από τον ε, Λετωνό συνάδελφο και άλλοι όμως έγραφαν αρνητικά. Άρα κάποιοι διαφωνούν. Να ολοκληρώσουμε λοιπόν τη συζήτηση και προηγουμένως πριν δώσω και πάλι το λόγο στον Τόμας Χέντελ επιτρέψτε μου να συνοψίσω κάποια ζητήματα που συζητήσαμε σήμερα το πρωί και ο Τόμας θα αναφερθεί σε αυτά που συζητήσαμε σήμερα το απόγευμα. Συζητήσαμε για την σύγκληση των ευρωπαϊκών οικονομιών και υπάρχει ευρεία συνένεση από αυτού. Οι οικονομίες μας πρέπει να συγκλίνουν, αυτό είναι το κλειδί στην επιτυχία της ε, ΟΝΕ μακροπρόθεσμα. Συζητήσαμε το επίπεδο αλληλεγγύης που χρειάζεται για να πετύχουμε αυτή τη σύγκληση ότι οι κανόνες πρέπει να βοηθούν αυτό το σκοπό και συζητήσαμε επίσης την ευθύνη, πιανού είναι η ευθύνη να τηρούνται οι κανόνες και αν υπάρχει συμμόρφωση. Συζητήσαμε επίσης για τον δημοκρατικό έλεγχο. Η έκθεση των πέντε πρόεδρων μας δίνει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβουμε. Αλλά θέτουν και νέα ερωτήματα και νέα διλήμματα. Όποιε προκλήσεις όμως πολιτικές και οικονομικές αντιμετωπίσουμε στο μέλλον, θα τις αντιμετωπίσουμε μαζί. Και το είπε ένας εκπρόσωπος. Αυτά τα πράγματα λύνονται από κοινού. Σήμερα αλλά και σε μελλοντικέ συζητήσεις θα έχουμε την ευκαιρία και την είχαμε και σήμερα να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει αμοιβαία κατανόηση. Και είμαι πεπισμένο ότι η ανταλλαγή απόψεων, όπω αυτή που είχαμε σήμερα, είναι ζωτική σημασία προκειμένου να πετύχουμε και την οικονομική σύγκληση αλλά και πολιτική σύγκληση. Πριν δώσω το λόγο λοιπόν στον συμπρόεδρό μου, τον κύριο Χάντελ, Πρώτα θέλω να τον ευχαριστήσω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μας φιλοξένησε εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πολύ και χειροκρέτημα για, από όλους εμάς για το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αγαπητοί συνάδελφοι, φτάσαμε στο τέλος της διακοινοβουλευτικής μας συνάντησης του 2016, τουλάχιστον το πρώτο τμήμα, επιτρέψτε μου να κάνω μερικές παρατηρήσεις. Δεν είναι δυνατόν να συνοψίσω σε λίγα λόγια αυτά που συζητήσαμε όλα. Αλλά ξέρετε είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης στο Κοινοβούλιο. Οπότε ίσως ε, να κάνω μερικές καταληκτικές παρατηρήσεις που νομίζω ότι είναι χρήσιμες για όλους μας. Ένα τέταρτο του ευρωπαϊκού πληθυσμού ζει στο ή κάτω από το όριο φτώχειας. Για μένα αυτό είναι ένα ζωτική σημασία θέμα που πρέπει να το συνδέσουμε με την πολιτική επενδύσεων. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε απόλυτοι στο διαχωρισμό μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων. Τις επενδύσεις που θα γίνουν μέσω του ΕΦΣΙ και του σχεδίου Juncker σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο θέλουμε να τις υποστηρίξουμε. Και κυρίως πρέπει να επικεντρωθούν στη δημιουργία απασχόλησης. Απασχόληση από την οποία να μπορεί κανείς να ζει αυτόνομα, χωρίς να χρειάζεται επιδόματα. Γιατί τα επιδόματα επίσης μετά από το δημόσιο κορβανά βγαίνουν και από τα ασφαλιστικά ταμεία. Πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε περισσότερο σε επενδύσεις που είναι προσαρμοσμένες στις ε, παρούσες και μελλοντικές ε, ανάγκες της αγοράς εργασίας. Έχουμε πολύ ψηλό επίπεδο κατάρτισης στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, ε, δυνατότητες πληροφορικής, δεξιότητες πληροφορικής. Οι επιστήμονες και οι επιχειρηματίες μας λένε ότι τώρα ξεκινάει η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και είναι ιδιαίτερα χρήσιμες αυτές οι δεξιότητες. Άρα πρέπει να κάνουμε κοινέ προσπάθειες και σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο ούτω ώστε να υπάρχουν αυτές οι δεξιότητες, να αυξηθεί το ποσοστό τους για να είναι απασχολήσιμοι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να βρουν θέσεις εργασίας και κάτι ακόμη. Και οι δύο ομιλήτριές μας έθεσαν το θέμα της γραφειοκρατίας και του κόστους της. Θέλω να τις παρακαλέσω να μην θεωρήσουν ως ε, γραφειοκρατικό άχθος να μην θεωρήσουν λοιπόν ότι τα δικαιώματα εργαζομένων τα νόμιμα δικαιώματα εργαζομένων να μην τα θεωρήσουν ως ε, γραφειοκρατικό κόστος γιατί σε πολλές χώρες επιτίθενται σε αυτά τα δικαιώματα στο όνομα της μείωσης της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα για παράδειγμα δεν είχε, δεν είχε ιδιαίτερη επιτυχία αυτή η προσπάθεια και θέλω να σας πω κάτι ακόμη ότι αν θέλουμε να οικοδομήσουμε τη μελλοντική Ευρώπη πρέπει να εστιάσουμε τις πολιτικές και οικονομικές προσπάθειές μας στην προσπάθεια να πείσουμε τους πολίτες για να επανέλθει η εμπιστοσύνη στην Ευρώπη. Γιατί όλο και λιγότεροι πιστεύουν στην Ευρώπη και όλο και λιγότεροι πιστεύουν γενικότερα στην δυνατότητα της πολιτικής να επηρεάσει τη ζωή τους και στη χειρότερη περίπτωση πιστεύουν όλο και λιγότεροι στις δυνατότητες της δημοκρατίας. Και εμείς λοιπόν θα τα ξαναπούμε στην Βρατισλάβα. Οι συνάδελφοι από τη Σλοβακία θα φιλοξενήσουν την επόμενη συνδιάσκεψη τον Οκτώβριο. Σας εύχομαι σε όλους καλή επάνωδο και ελπίζω οι συζητήσεις μας αυτό το διήμερο να σας ωφέλησαν. και ευχαριστώ πολύ.